Buongiorno, colleghe, e colleghi. Καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Invito tutti a prendere... Παρακαλώ καθίστε όλοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Για μια ακόμη φορά σας καλημερίζω. Έχω λάβει από τις πολιτικές ομάδες και από τους μη εγγεγραμμένους τους ορισμούς στις κοινοβουλευτικές επιτροπές επί τη βάση του άρθρου 209 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κατάλογος των ονομάτων για τη σύνθεση των επιτροπών έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας καλούμεθα να εκλέξουμε τους κοσμήτορες σήμερα. Έχω λάβει τις εξής υποψηφιότητες. Κυρία Μπένοβα, ο κύριος Μπουαγιέ, ο κύριος Κάζα, ο κύριος Κάσκι και η κυρία Σάντερ. Οι υποψήφοι δέχονται τις υποψηφιότητες αυτές Ο αριθμός των υποψηφίων δεν ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων που πρέπει ε, να καλύψουμε και γι' αυτό επί τη βάση του άρθρου 15 παράγραφος 1 διαβοή τους εκλέουμε. E ε, Καλώς λοιπόν. Vi sono, vi sono, vi sono, devo Έχουν, ε, έχει ζητηθεί από κάποιον η μυστική ψηφοφορία. Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Συνεπώς λοιπόν οι υποψήφοι ε, έγιναν πλέον κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχαίρω τους συναδέλφους για την εκλογή τους. Però una votazione la dobbiamo fare, come sapete. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία. Με την σειρά, πρέπει να καθορίσουμε τη σειρά για την απόδοση των ψήφων για τους πέντε υποψήφιους κοσμήτορες. Περνάμε λοιπόν σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των κοσμητόρων. Πολλοί από εσά έχουν ήδη προπονηθεί ε, για στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μυστική ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μία δοκιμή. Ας κάνουμε μία επιπλέον δοκιμή όπως αυτή που κάναμε χτες με ονόματα τραγουδιστών, όχι πραγματικών βουλευτών για να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Στις οθόνες σας θα έρθουν κάποια ονόματα πάρα πολύ γνωστά και μπορείτε εσείς με το βελάκι να διαλέξετε ακριβώς τα ονόματα που επιθυμείτε. Αυτό θα το κάνετε τη στιγμή που ξεκινήσει η ψηφοφορία, έτσι ώστε να καθορίσετε τη σειρά. Λοιπόν, ας κάνουμε τη δοκιμή την οποία είπα. Ψηφίσατε όλοι. Παρακαλώ να ψηφίσετε, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος παρακαλώ να ψηφίσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε. Κάναμε και χτες μια τέτοια δοκιμή, αλλά πρέπει να ψηφίσετε όλοι. Πρέπει να ψηφίσετε στη συγκεκριμένη περίπτωση 5 εκ των 8. Πέντε ονόματα από τα 8 τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη σας. τουλάχιστον για τρεις, ε, τρία ονόματα πρέπει να ψηφίσετε, αλλιώς δεν θα θεωρηθεί ε, έγκυρη η ψήφο σας. Λοιπόν, παρακαλώ να προχωρήσουμε να επιλέξετε τα ονόματα τα οποία επιθυμείτε. Άρχεται η συνεδρίαση. Ψηφίσατε όλοι. Επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος αν ψηφίσατε όλοι. La votazione Πέρα της ψηφοφορίας. Ψηφίσαντες 559. Λευκή Άκυρη 86 έγκυρες ψήφοι 473. Λοιπόν, έχουν εκλεγεί δηλαδή οι τραγουδιστές τους οποίους επιλέξατε. Λοιπόν, δούλεψε το σύστημα, η δοκιμή έγινε, ας περάσουμε τώρα πια στην κανονική ψηφοφορία για τους κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να καθορίσουμε ακριβώς την σειρά με την οποία θα εκλεγούν. Έχουμε πέντε θέσεις, θα πρέπει τουλάχιστον τρεις να ψηφίσετε γιατί αλλιώς η ψήφο σας θα θεωρηθεί άκυρη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Επαναλαμβάνει τώρα ο Πρόεδρος αν έχετε όλοι ψηφίσει. Έχετε όλοι ψηφίσει. πέρα της ψηφοφορίας. Ψηφίσαντες 574. Λευκές και άκυροι 71. Έγκυρες ψήφοι 503. 407 ψήφοι, Ιαν Σάντερ, Στη δεύτερη θέση η κυρία Μπένοβα 391 ψήφοι. Con gli stessi voti 390... Με τον ίδιο αριθμό ο κύριος Κάζα 391 ψήφοι. 317 ψήφοι για τον κύριο Ζήλ. με 261 ψηφίο ο κύριος Κάσκι. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο, συγχαίρω τους νέους κοσμήτορες με βάση το 18 έχει καθοριστεί πλέον η σειρά μέσω της ψηφοφορίας που μόλις έγινε. Θα ανακοινωθεί επίσημα στους προέδρους των οργάνων, το αποτέλεσμα στους ε, προέδρους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κλείσαμε προς το παρόν και ξεκινάμε πάλι στις 10.30. Με βάση το άρθρο 18 η σειρά των κοσμητόρων καθορίζεται από τη σειρά με την οποία εκλέγονται και στην περίπτωση ισοψηφίας από την ηλικία.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 Παρακαλώ τους συναδέλφους να πάρουν θέση. Κυρίσουμε την ε, επανάληψη της Συνόδου. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 20 και 21 Ιουνίου. Να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στον πρόεδρο Τούσκ, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Παρακαλώ, πρόεδρε, έχετε το λόγο. Να καλημερίσω και τον Επίτροπο σέφκοβιτς που είναι μαζί μας. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι αγαπητή Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον εκλεγέντα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή τύχη και ευελπιστώ σε αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί την αγνήσια, αυθεντική Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, γιατί τα μέλη εκλέγονται με άμεση για καθολική ψηφοφορία. Ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει την σημαντική ε, δημοκρατική νομοποίηση των ηγετών. Ε, και τα δύο θεσμικά όργανα είναι δημοκρατικά. Και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την Ευρώπη. Και γι' αυτό πριν την πρόταση που κάναμε για τις ηγετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συναντήθηκα με κροσόπους σας πολλές φορές. Και αυτό το έκανα όχι μόνο από σεβασμό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για να διασφαλίσω ε, σωστή διαδικασία αποφάσεων και διαφανή. Και μάλιστα καταφέραμε έγκαιρα να λάβουμε τις αποφάσεις και μάλιστα και σχετικά πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι θετικές. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε δύο γυναίκες και δύο άνδρες για να ηγηθούν ε, σημαντικών αξιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που υλοποίησαμε μια τέλεια εκπροσώπηση των ε, φίλων σε ηθήνουσες θέσεις. Αυτή είναι μια πολύ θετική αλλαγή. Ευρώπη δεν μιλάει απλώς στη θεωρία για τις γυναίκες, αλλά επιλέγει γυναίκες. Και ελπίζω αυτή η επιλογή να εμπνεύσει πολλές γυναίκες και κορίτσια να δώσουν τη μάχη για τα πάθη τους ε, και τις πεπιθήσεις τους και να εμπνεύσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μελλοντικές αποφάσεις του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, στη διάρκεια της επιλογής των υποψηφίων είχα στενές επαφές με τους ηγέτες των Πρασίνων, κυρίως με τη Σκακέλερ και τον Φιλίπ Λάμπερτ. Και πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία με τους πράσινους και η παρουσία τους στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα βοηθήσει όχι μόνο τις κυβερνητικές ε, συμμαχίες και συνασπισμούς, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς όλους τους εταίρους να συμπεριλάβουν και τους πράσινους ε, στις ε, διάφορες διαδικασίες, παρόλο που δεν ε, έχουν ακόμη κάποιον από τους πράσινους. Και ελπίζω η der Leyen να ακούσει αυτό το μήνυμα και αυτή την έκκληση, αν και θα της το διαβιβάσω και προσωπικά αυτό το μήνυμα. Και όπως ξέρετε, σε πολλές χώρες η πράσινη είναι το σύμβολο της ε, ελπίδας και της ελευθερίας και πιστεύω σε αυτό το συμβολισμό. Και σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές ευαισθησίες στην Ευρώπη, θα ήθελα να αναφέρω την ενότητα και τη γεωγραφική ισορροπία. Όπως ξέρετε, προσωπικά έδωσα μάχη να διασφαλίσω την ευρωπαϊκή ενότητα στο παρελθόν. Ε, δείχνοντας ελεγγύη προς την Ουκρανία, βοήθεια προς την Ελλάδα, ε, στη, στη μεταναστευτική κρίση. Και μερικές φορές επιτύχαμε περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, ενώ ταυτόχρονα καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι. Και Γι' αυτό, και αυτό γιατί οι ηγέτες ε, έχουν επίγνωση της ισχύω που έχει η ενότητα. Και σίγουρα είναι σαφές ότι μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να αντισταθμίσουμε, να είμαστε το αντίβαρο των πιο ισχυρών παγκόσμιων εταίρων μας. Στην τελευταία διάσκεψη κορυφής καταφέραμε να καταλήξουμε και σε κάποιες ε, συνενετικές ε, αποφάσεις. Χρειαστήκαμε τρει μέρε γι' αυτό, αλλά θέλαμε όλε οι χώρε, μεγάλε και μικρέ από κάθε πλευρά τη Ευρώπη, να συμμετέχουν στην επιλογή των ηγετικών θέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωση σε ό,τι αφορά του εκπροσώπου τη Ανατολική Ευρώπη στο γενικό οικοδόμημα και το οργανόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα κάποιοι πρωθυπουργοί από τη σοσιαλιστική οικογένεια ε, έδωσαν έκαναν δεσμεύσει για τη γεωγραφική ισορροπία και εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλυψε και κάποια άλλα θέματα, αλλά όπως ξέρετε ε, έχουμε δώσει τα συμπεράσματά μας, είναι γνωστά, γι' αυτό δεν θα ήθελα να γρηγορήσω και να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι και πάλι καλή τύχη. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Τούς και τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίτροπε Σεύστοβιτς, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αξιότιμοι βουλευτές. Έχω την χαρά και την τιμή να απευθυνθώ εξ ονόματος του Πρόεδρου Γιούνκερ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, πρώτη συνεδρίαση της νέας θετίας. Συζητήσαμε τα θέματα των θέσεων απασχόλησης, των θέματα μάλλον των θέσεων και των ε, ονομάτων που θα ε, έχουμε στην Ευρώπη νυχθημερών, γιατί συχνά παίρνει χρόνο το να βρούμε τους σωστούς συμβιβασμού και αξίζει να βάλουμε τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση όταν μιλάμε για θέσεις εξουσίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια και γι' αυτό είμαι χαρούμενος, ευτυχής που ε, το Κοινοβούλιο ε, εξέλεξε τον πρόεδρο Σασόλη για την ενδεχομένω πιο δύσκολη δουλειά από όλε. Στα τελικά, ο κύριος Σάκοβιτς, σας συγχαίρω λοιπόν κύριε πρόεδρε και συγχαρητήρια σε όλους τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, εκλογή τους. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όχι μόνο εξ ονόματος προσωπικό, αλλά και εξ ονόματος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των συναδέλφων στο Σώμα των Επιτροπών. Να υπογραμμίσω ότι όλοι προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλους σας. Το ίδιο ισχύει και όλους, για όλους τους υποψηφίους που έχουν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσολαν Leyen, που έχει πραγματικά ό,τι χρειάζεται για να ηγηθεί το θεσμικό μας οργάνος. Φυσικά το Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία κουβέντα και θα το συζητήσουμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αφορούσε μόνο ε, τις θέσεις αυτές και οι διάφορες προσωπικότητες. Το θέμα ήταν και οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για τα επόμενα πέντε έτη και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολλο, πολλά κοινά σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα. Να τονίσω δύο μόνο ζητήματα. Καταρχάς την κοινωνική διάσταση. Σήμερα πιο πολύ από ποτέ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος έχει ευκαιρίες. Μια εποχή που οι Ευρωπαίοι έχουν μεγάλες προκλήσεις και περνούν διάφορες μεταβάσεις, οικονομικές, οικολογικές, ψηφιακές μεταβάσεις. Όλα αυτά έχουν σημαντικό αντικτύπο στην καθημερινή ζωή. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να τονίσω και πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό, το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ήταν πραγματικά η πιο περήφανη στιγμή μου ως επίτροπος, όταν είχα την τιμή και προσυπέγραψα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που κατά πάσα πιθανότητα ήταν η πιο σημαντική συμφωνία στις πρόσφατους καιρούς ε, στη Νέα Υόρκη, τη, η Συμφωνία των Παρισίων. Ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εργαστήκαμε όλοι πάρα πολύ σκληρά και συνεργαστήκαμε πολύ σκληρά μαζί σα για να μπορέσουμε να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων και των δεσμεύσεων που είχαμε αναλάβει. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι είμαστε η πραγματική οικονομία που έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι και 40% ε, σε σχέση με το επίπεδο του 90 μέχρι το 2030. Και ξέρουμε ότι η σκληρή αυτή η εργασία θέτει τις βάσεις για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μέχρι το 2030. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι η πιο φιλόδοξη αυτή στοχοθεσία Μεγάλε οικονομίε και έχουμε και το νομοθετικό πλαίσιο πλέον για να τα απεξέλθουμε στι δεσμεύσει μας αυτές. Για να συνεχίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγείται όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να... να τα λόγια να έρθουν και οι πράξει σε ό,τι αφορά το 2030. Αλλά η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να σταματήσει το 2030. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, στην Ευρώπη να δεσμευτούμε την οδό της ε, κλιματικής ουδετερότητας ε, σε ό,τι αφορά το 2040, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένας ε, καθαρός πλανήτης για όλους είναι προς το συμφέρον μας, όλων μας, όχι μόνο το οικονομικό μας συμφέρον, αλλά αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και κάποια λίγα κράτη-μέλη που θα πρέπει να επιταχύνουν Γι' αυτό λοιπόν ε, έχουμε αφιερώσει, αφιερώσει 25% του προϋπολογισμού σε τέτοιους σκοπούς και έχουμε ξεκινήσει και μια βιώσιμη στρατηγική χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν και τα ιδιωτικές επενδύσεις να στραφούν σε πιο βιώσιμες οδούς. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά, εκτός και αν έχουμε το σωστή χρηματοδότηση τη σωστή στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένω ότι θα πρέπει να πετύχουμε και μία συμφωνία για το μελλοντικό πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Το φθινόπωρο μάλιστα. Και υπολογίζω σε εσά, αξιότιμοι βουλευτέ, ότι θα είναι δική σα προτεραιότητα να ολοκληρώσετε τι διαπραγματεύσει με τη Φιλανδική Προεδρία το εκλογικό κοινό ευρωεκλογέ είναι σαν μια αποτελεσματική Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά, αποτελεσματικά. Και ξέρουμε ότι αυτό θα το πατήχουμε μόνο αν ολοκληρωθεί ο προπολογισμό, το σχέδιο προπολογισμού εγκαίρω. Αυτό χρειάζεται αποφασιστικότητα. Έχουμε 100.000 ε, ε, προγράμματα συνοχής, ερευνητές, ε, φοιτητές, εράσμους. Κάθε μέρα μετράει αν θέλουμε να ξεκινήσουν όλα αυτά τα προγράμματα από 1η Πρώτου του 2021. Εδώ πραγματικά όντω ο χρόνος είναι χρήμα. Και ελεκτικά, και μιας και μιλάμε για χρήματα, να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπιστώσαμε πως η σκληρή εργασία μας για την εμπάθυνση, την οικονομική και την νομισματική απέδωσε καρπούς. Έχουμε ένα σταθερό νομίμισμα σήμερα με πληθωρισμό 1,8% στην Ευρωζώνη. Οι ευρωπαϊκέ τράπεζε είναι πιο ασφαλεί, πολύ πιο ασφαλεί από ό,τι πριν την ε, οικονομική κρίση και ε, το buffer είναι περίπου στο 20% των συνολικών δαπανών σε σχέση με το 10% πριν από την κρίση. Και ω αποτέλεσμα η Τραπεζική Ένωση και τα κόκκινα δάνεια, τα μη των δάνεια, φτάνουμε στο επίπεδο σχεδόν προκρίσης. Αλλά δεν μπορούμε να επανεπαυθούμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα για να πετύχουμε πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, τα ε, εργαλεία για την σύγκληση, για την ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικά εργαλεία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση και σωστή διακυβέρνηση των εργαλείων αυτών. Επίση, χρειάζονται πιο πολλέ προσπάθειε για την ε, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα να είναι αξιόπιστο να είναι έγκυρο. Να ενταχθεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε βάθος χρόνου και επίσης στην κοινή εγγύηση ε, αποταμιεύσεων καταθέσεων για να μην μας χτυπήσει η επόμενη κρίση πρωτού έχουμε προετοιμαστεί για τέτοια θέματα. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε ακόμα και είμαι λοιπόν ευτυχή που με την ολομέλεια αυτή ξεκινούν οι δικέ σα εργασίε. Είναι μόνο η αρχή αξιότιμοι βουλευτέ. Επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο-τρία λόγια για τα άλλα θέματα τα οποία συζητήσαμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταρχά, να επαναλάβω την πλήρη υποστήριξή μα για την Κύπρο σε ό,τι αφορά τι ε, συνεχιζόμενε δραστηριότητε παράνομε τη Τουρκία για εξόριξη. Στο ΣΥΠΙΟ είχαμε διευκρινίσει και πει ο πρόεδρο Γιούγκερ ότι σε αυτό το θέμα είναι Κύπριο και είμαι πεπισμένο ότι ε, στο Συμβούλιο αυτό όλοι Όλα τα κράτη-μέλη είπαν ότι είμαστε Κύπροι σε αυτό το θέμα. Σε πνεύμα αλληλεγγύη, λοιπόν, εργαζόμαστε για συγκεκριμένε δράσει και αναζητούμε συγκεκριμένε ενέργειε. Και διαβεβαιώ τον λαό τη Κύπρου ότι θα επιδείξει η Ευρώπη αλληλεγγύη προ την Κύπρο και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Δεν μπορώ να, να απευθυνθώ στην Κύπρο χωρί να απευθύνω τα συλληπιτήριά μου προ την οικογένεια του Δημήτρη Χριστόφια και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αξιόπιστη ε, πρόπτικη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή. Είναι νομίζω η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για να υπάρξει σταθερότητα, να ξεπεραστούν τα διμερή θέματα και να συνεχιστεί και αυτή η τάση μεταρρύθμισης που πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς. Τα ένα απόφαση για τις ε, έναξη διαπραγματεύσεων μέχρι τον Οκτώβριο για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Και η Επιτροπή θέλει να κάνει ανοιχτέ συζητήσει ε, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ, είναι βασικό οι δύο αυτέ χώρε και όλη η περιοχή να συνεχίσουν τι μεταρρυθμίσει. Οι μεταρρυθμίσει αυτέ, οι προσπάθειε αυτέ γίνονται βασικά για του πολίτε της χώρας, των χωρών αυτών και της περιοχής αυτής για να υπάρξει δικαιοσύνη, να υπάρξει κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Και τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω την πλήρη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία μετά από τα θέματα στην ανατολική πλευρά της χώρας. Ε, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία του Μίνσκ θα, οι συμφωνίες του Μίνσκ θα τηρηθούν απόλυτα την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενή σύνοδο θα συζητήσουμε όλα αυτά και θα κάνω προσωπικά ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα συνεχιστούν η, μεταβάση, η διαμετακόμιση αερίου μέσω της Ουκρανίας στην επόμενη περίοδο. Και να σας ενημερώσω επίσης ότι οι επόμενες τριμερείς συμφωνίες μεταξύ Επιτροπής ε, Ρωσίας και ε, Μίνσκ θα ξαναξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτ. Και τώρα ο λόγο στον Πρόεδρο Γκονζάλε Πόν, εκ του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Θα ήθελα εκ μέρου του μεγαλύτερου κόμματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγχαρώ τον Πρόεδρο σα όλοι και να το ευχηθώ καλή τύχη. Σας ψηφίσαμε, κύριε Πρόεδρε, μην το ξεχνάτε ούτε τώρα ούτε μετά από δυόμιση χρόνια. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ταγιάννη που ανέκαθεν υπεράσπισε την τιμή και την αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του. Επίση, θα ήθελα να συγχαρώ του συναδέλφου, του νεοεκλεγέντε και του πιο παλέμαχου, γιατί εμεί θα πρέπει να υπομιστούμε την ευθύνη να εκπροσωπήσουμε τον ευρωπαϊκό λαό. Είμαστε το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τον Ευρωπαϊκό Λαό. Δεν θα συγχαρώ όμω το Συμβούλιο, με όλο το σεβασμό που τρέφω προς τον πρόεδρο Τούσκ. Πραγματικά δεν μπορείτε να είστε υπερήφανοι για αυτό που κάνετε, για τον τρόπο που δράσετε, είτε για το βέτο, είτε για την έλλειψη σεβασμού που δείξατε στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα στους ε, ε, εξτρεμιστές, ε, δεν ξέρω αν είναι παρόντες, που την περασμένη Τρίτη γύρισαν την πλάτη στον ύμνο της Ευρώπης. Θα ήθελα να πω ότι εμείς ποτέ δεν θα γυρίσουμε την πλάτη στον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν αρχές και εκείνων που δεν έχουν. Σήμερα λαμβάνω το λόγο εκ μέρου μια πολιτική ομάδα που είναι βαθύτατα φιλοευρωπαϊκή, που συνέβαλε στην διαμόρφωση της Ευρώπη από τα θεμέλια τη Είμαστε ε, μια ομάδα ε, από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ομάδα που σε αντίθεση με άλλες είναι έτοιμη να κάνει θυσίες ε, και υποχωρήσεις για να καταλήξει συμφωνίες. Είμαστε μια ομάδα που είμαστε περήφανοι για τον candidate μας, τον κορυφαίο μας υποψήφιο στις πρόσφατες ευρωεκλογέ, τον Μάνφρεντ Πέμπερ. Μάνφρεντ, έχει την απόλυτη υποστήριξή μας, γιατί ε, πραγματικά σήμερα ενσαρκώνει το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας απέναντι στο Συμβούλιο η Ευρώπη, εκτό ότι φαίνεται δημοκρατική, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και δημοκρατική. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εδώ και χρόνια υπέρ τη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου, του Spitzenkandidat. Γιατί πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίζουν για αυτόν που τους κυβερνά, αλλά και ποιος τους κυβερνά. Επίσης διαβεβαιώ αυτή την πενταετία θα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στις κάλπες και όχι στις κλειστές πόρτες. Και μάλιστα μπορεί να είναι νομοποιημένες οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να επιβάλλονται με την ισχύ του κράτους στην θέληση των Ευρωπαίων πολιτών που εκπροσωπούνται στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το ΕΛΚ, θα υποστηρίξει την υποψήφια που πρότεινε το Συμβούλιο από υπευθυνότητα και μόνο γιατί ανήκει στην πολιτική οικογένεια που κέρδισε τις ευρωεκλογέ. και ε, θέλουμε ε, μία ικανή υποψήφια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μάχη για τα συμφέροντα της Ευρώπης. Και ως πολιτική ομάδα είμαστε υπερήφανοι που η Ούρσουλα Βαντελέιεν θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και Χαιρόμαστε που είναι μια γυναίκα που ανήκει στην κεντροδεξιά πολιτική παράταξη. Βέβαια, το Συμβούλιο και η υποψήφια του θα πρέπει να διαπραγματευτούν το πολιτικό του πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στα μέλη του Συμβουλίου θέλουμε να ζητήσουμε να κάνουμε ε, συζητήσεις και να σταματήσουμε ε, με μυστικές ε, συνωμοσίε και πίσω από κλειστές πόρτες να αποφασίζουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία του and Candidate» δεν αφορά μια γυναίκα ή έναν άνδρα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να διαλέγουν ποιο θα του κυβερνά στην Ευρώπη. Αυτό είναι πραγματικά μια επαναστατική ιδέα που φέρει το όνομα Δημοκρατία. Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποψήφιο για τη θέση του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει. Αλλά το Συμβούλιο δεν δικαιούται να αγνοεί του υποψηφίου ε, που ε, ψήφισαν ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι πολίτε. Κύριε Τούσκ, ε, πραγματικά δημιουργήσατε μια ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγνοεί την ε, Ανατολική Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος από την Ανατολική Ευρώπη. Και κύριε Τούσκ, ασκήσατε βέτο σε, στον υποψήφιο που ψήφισαν 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ισοδυναμεί με τον πληθυσμό της πατρίδας σας και της δικής μου. Βάλατε βέτο για αυτόν τον άνθρωπο και προτείνατε υποψήφια της, ε, ε, της, της Προεδρής Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ενώ είχαμε πόσες αντιπροεδρίες ακόμη θα ε, δεχτείτε πέραν της Προέδρου ε, χωρίς διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς θα πείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποιο θα ορίσει πρόεδρό του. Για... Ε, και επίσης για πόσο χρόνο θα κάνουμε τη μοιρασιά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ε, εσείς ορίσατε επίσης ε, τη, την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν να ήταν ένα πολιτικό στόχο. Αυτό είναι πραγματικά πολύ κακή δημοκρατική κουλτούρα, μια πολύ κακή δημοκρατική διαγωγή. Ουσιαστικά παίξατε το παιχνίδι των ευρωσκεπτικιστών και των εθνικιστών. Κανένα από του προέδρους, ε, του που συμμετέχουν στο Συμβούλιο δεν θα τολμούσε να κάνουν αυτά που έκαναν στο Συμβούλιο ε, στις πατρίδες τους, γιατί θα του εμπόδιζε το Συνταγματικό Δικαστήριο. Και πραγματικά έχετε τύχει που το άρθρο 7 της ε, συνθήκη τη Λισαβόνα, δεν ισχύει για το Συμβούλιο. Γιατί πραγματικά σήμερα θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Γιατί ανοίξατε μια πολύ σοβαρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποιο αποφασίζει την Ευρώπη. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Η κοινοβουλευτική ομάδα δική μου πιστεύει ότι στην Ευρώπη ο λαός θα πρέπει να αποφασίζει, γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Γκονζάλε Πόνς. Και τώρα η πρόεδρος Γκαρσία Πέρες. E Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Στις ε, ευρωεκλογέ του Μαΐου, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, μας διαμήνυσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πιστεύουν στην Ευρώπη, έχουν εμπιστοσύνη, αλλά θέλουν αλλαγέ. Και σα διαβεβαιώ ότι η δική μου πολιτική ομάδα έχει τη δέσμευση και την ευθύνη να προωθήσει αυτέ τι αλλαγέ. Και νομίζω ε, αναφυσβήτητα ο καλύτερος ε, ε, ηγέτης αυτών των αλλαγών θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Φραντς Τίμερμανς, γιατί θα είχαμε και ένα speech and candidate που θα είχε την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις δημοκρατικές μας αξίες και αρχές. Και δεύτερον, κάτι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ο δικός μας υποψήφιος ε, παραγωνίστηκε γιατί ήταν υπέρμαχος του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών. Και είναι προφανές ότι εμείς θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές και οι αξίες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό στην πολιτική που επίση έχει θεμελιώδη σημασία. Η συνέπεια. Και δεν είναι συνεπές να έρχεστε εδώ και να μας προτείνετε ε, αυτή την ε, απόφαση του Συμβουλίου ε, και να λέτε ότι θα υπερψηφίζετε. Απ' τη μια μάλλον την ρίχνετε στα σκουπίδια και απ' την άλλη λέτε ότι θα υπερψηφιστεί. Δεν είστε συνεπείς. Η πρωταρχική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αν είμαστε συνεπείς με αυτές τις αρχές, ήδη εδώ και πολύ καιρό θα είμαστε πολύ πιο συντονισμένοι και κατηγορηματικοί για να μιλούμε για πολιτική στην Ευρώπη. Για να μιλούμε για το πώς είμαστε ικανοί να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να φροντίσουμε ώστε να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική και για το πώς η πολιτική μας ομάδα θα ηγηθεί των πολιτικών αλλαγών στην Ευρώπη. Χαίρομαι που τα Ιταλικά δικαστήρια απελευθέρωσαν την καπετάνιο, την Καρόλα Ρακέτε. Αυτό συμβαίνει γιατί πραγματικά υπάρχει διάκριση εξουσιών. Μόνο με διάκριση εξουσιών γίνεται δυνατό κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό έχει ζωτική σημασία να διαφυλάξουμε αυτή τη διάκριση εξουσιών απέναντι ε, στους ε, ε, όσους θέλουν να την υποσκάψουν. Επίσης, έχουμε δραματικές αλλαγές λόγω της έλλειψης αλληλεγγύης. Είναι πραγματικά ανέντιμο να ποινικοποιούμε αυτούς που σώζουν ζωές και να καρπονόμαστε πολιτικά την δυστυχία αυτών των ανθρώπων. Και αφού μιλούμε για πολιτική και περιεχόμενο, δεν θα στηρίξουμε καμία υποψήφιο και κανέναν υποψήφιο που θα προτιμήσει την ακινησία απέναντι στην ανάγκη των αλλαγών σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, θέλουμε την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και την οικολογική μετάβαση. Ο χρόνος δεν περιμένει, το ρολόι δεν ε, περιμένει. Μας το λένε αυτό οι έφηβοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατεπίγουσα η κατάσταση στις κλιματικές αλλαγές. Μας το λένε οι έφηβοι, οι νέοι. Ας μη τους απογοητεύσουμε. Γι' αυτό θα είμαστε πολύ απαιτητικοί με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής. Οι κλιματικές αλλαγές χρειάζονται πραγματικά μεταρρύθμιση με δίκαιη μετάβαση και βιωσιμότητα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες. Θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις των Παρισίων Εμεί ήμασταν ανέκαθεν πρωτοπόροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε πλειοψηφίε ώστε να παροτρύνουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να συγχαρώ τη Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου για τι προτάσει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον που έκανε. Συνεχίζουμε να μιλούμε για πολιτική. Θέλουμε ένα πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα είναι φιλόδοξο για να υλοποιήσουμε τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα επιτεύγματα με λιγότερου πόρου. Γι' αυτό και θα δώσουμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε τι πολιτικέ μα. Θυμάστε την Ευρώπη 2020. Δεν καταφέραμε, ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της, να υλοποιήσουμε τους στόχους. Έχουμε 5 ε, εκατομμύρια μόνο από τα 20 που θέλαμε να ξεφύγουν από την φτώχεια. Και άλλοι ε, εσφετερίζονται και αξιοποιούν την κρίση, ενώ άλλοι πληρώνουν τα σπασμένα. Δεν μα αρκούν ε, τα μεγάλα νούμερα. Μα ενδιαφέρει ο άνθρωπο και θέλουμε η οικονομική ανάπτυξη να φτάνει στου Ευρωπαίου πολίτε, στου άνδρε και τι γυναίκε τη Ευρώπη, που θα πρέπει να ζουν καλύτερα, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Θέλουμε μια αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ώστε να περιλαμβάνει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τον κοινωνικό πυλώνα, των κοινωνικών δικαιωμάτων δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την, την ε, νομισματική ένωση. Ας μην περιμένουμε μια καινούργια κρίση για να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωζώνη, για να έχουμε προπολογισμό τη Ευρωζώνη και μία εγγύηση των καταθέσεων. Για να υλοποιήσουμε όμω αυτού του στόχου, θα πρέπει ταυτόχρονα να επεξεργαστούμε και ένα γενικό πρόγραμμα. Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη παγκοσμίω, να προωθήσουμε ανθρω... προδιαγραφέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικέ προδιαγραφέ περιβαλλοντικέ στι πολυμερεί μα συμφωνίε. Οι πολίτε περιμένουν περισσότερα από εμά. Θέλουν να προασπίσουμε τα κοινωνικά και εκτιμένα, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα, τα δικαιώματα τη κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, η Επίση, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αδικίε, όπω είναι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά στα χέρια μας, στο χέρι μα είναι να σταματήσει επιτέλους η βία λόγω φύλων, να σταματήσει οι γυναικοκτονίες ε, και η βία κατά των γυναικών μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις από τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και να χρονοτριβούμε. Είμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη βάσει των αξιών της ισότητας, της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης. Και θα συνεργαστούμε με όσους προασπίζονται αυτούς τους στόχους. Ας μην απογοητεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πέρες, ε, κυρία Πέρες, ε, ο κύριος Σόλος, ο πρόεδρος Σόλος, για την ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που εξελέγησαν στα ηγετικά αξιώματα του Κοινοβουλίου και σας τον ίδιο. Μαζί σας και με τη νέα μας ομάδα, με την ομάδα Renew Europe, θα κοιτάξουμε να γίνει ακόμη πιο ηχηρή η φωνή του Κοινοβουλίου και να ακουστεί παντού. Αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστω είναι να υπάρξει μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό τη διαδικασία για τον ε, ορισμό των ε, πρώτων αξιωμάτων που θα αναλάβουν πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να συζητάμε ονόματα, γεωγραφική ισορροπία, την ισορροπία των φύλων, αλλά όσο δεν είναι δημοκρατική και διαφανή η διαδικασία για την επιλογή των προσώπων που ηγούνται στην Ευρώπη, δεν θα έχουμε πετύχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οι συνάδελφοι που μίλησαν προηγουμένως εξέφρασαν κάποιες απόψεις και είπαν τη γνώμη τους για το πώς εξελέγησαν αυτοί οι άνθρωποι. Πρόεδρε, δεν υπάρχει ακόμη ισορροπία. Δεν υπάρχει γεωγραφική ισορροπία. Η Ανατολική Ευρώπη δεν εκπροσωπείται όπως εκπροσωπείτε όταν εσείς ε, οριστήκατε, διοριστήκατε μάλλον στο αξίωμα που ακόμα κατέχετε. Χρειάζεται λοιπόν ε, μια διαδικασία που να λαμβάνει υπόψη όλες τι διατάξει τη Ευρωπαϊκή συνθήκης και μια διαδικασία εντελώς δημοκρατική. Κυρίες και κύριοι του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αν πραγματικά θέλετε να λέγεστε δημοκράτες, να διέπεστε από δημοκρατικό πνεύμα, εάν θέλετε ε, όσοι καταλαμβάνονται σε ηγετικέ θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρείται ότι πραγματικά εκπροσωπούν του πολίτε, θα πρέπει να υπάρχουν και ε, διακρατικά, διασυνοριακά ψηφοδέλτια. Οι ε, εκλεγμένοι να εκλέγονται από όλου του πολίτε ταυτόχρονα, όχι μόνο από Γερμανού, Ισπανού, Ολλανδού ξεχωριστά η διαδικασία των Spitzenkandidaten να ε, είναι επιλογή όλων των Ευρωπαίων πολιτών ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν να προτείνουμε και αυτό είναι μια αλλαγή του Ευρωκοινοβουλίου. Να μην περιμένουμε πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν ε, αυτό που θα ήταν ε, κανονικά δική μας αρμοδιότητα. Αυτό λοιπόν προτείνει η δική μας ομάδα, η New Europe, είναι μια μια ευρωπαϊκή διάσκεψη ε, για τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας των εκλογών ή μια συνέλευση με διάρκεια διετή ε, μια συνέλευση ε, που θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ενώσεων των πολιτών, για να βελτιώσουμε τι διαδικασίε που αυτή τη στιγμή ισχύουν. Κυρία Γκονζάλε Πον, συμφωνώ απολύτω. Κυρία ε, Γκαρσία Περέ, επίση συμφωνώ. Χρειαζόμαστε κόσμο που πραγματικά να εκπροσωπεί του πολίτε, του Ευρωπαίου πολίτε. Αλλά ας κοιτάξουμε πρώτα να καθορίσουμε τη σωστή διαδικασία και να υπάρξει πραγματικά ανταλλαγή απόψεων, όχι τελευταία στιγμή, όταν το Συμβούλιο έχει λάβει, λάβει τι αποφάσει του. Α εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διάρκεια αυτή τη θητεία, ώστε στι επόμενε εκλογέ να μην ζήσουμε τα ίδια. Να υπάρξει διαδικασία που να συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, τα κάτι μελη και να μην χάνουμε χρόνο ανταλλάσσοντα ε, ε, δημιουργίες και τοποθετήσεις δρυμίες. Ε, αυτό υποστηρίζω εγώ, αυτό προτείνω και ελπίζω να σας βρω σύμφωνος. Έχουμε χρόνο στις επόμενες ευρωεκλογέ για να καταρτιστεί μια τέτοια διαδικασία. Κατά δεύτερον, οι ευρωπαϊκές αξίες, ε, δηλαδή το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Και βεβαίως αυτό θα πει κιόλα ε, δημοκρατία. Ε, είναι σημαντικό σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να ορίσουμε μια σειρά από αρχές για την προστασία του κάτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα μηχανισμό κυρώσεων που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Έναν μηχανισμό πρόληψης που θα δείχνει σε κάθε κράτο μέλο ποια είναι τα όρια εντό των οποίων μπορεί να κινηθεί. Τι γίνεται όταν παραβιάζει του κανόνε για το κράτο δικαίου και για τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει σύντομα να διορίσουμε και τον υπεύθυνο για την ε, εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και αυτή αυτό το λειτουργήμα πρέπει να καλυφθεί από κάποιον πολύ γρήγορα για να περάσει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εδώ μόνο για να τιμωρεί ε, έχει ρόλο και να προλαμβάνει και έχει τον τρόπο να το κάνει. Κατά τρίτον, χρειαζόμαστε και ένα νέο όραμα. Ένα πολιτικό όραμα για τα θέματα του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά ε, και θα πρέπει για τις κλιματικές αλλαγές να φροντίσουμε να υπάρξει και κάποια ε, παράλληλη εξέταση και σύγκληση με τους ε, οικονομικούς και κοινωνικούς μας στόχους ε, στην Επιτροπή. Είναι γνωστό πόσες φορές έχει τοποθετηθεί σχετικά με αυτά το Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως τώρα να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ατζέντα. Αυτό που έχει ήδη κάνει το Συμβούλιο για το 2019-2024 είναι ήδη ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο να εργαστούμε εντατικά σε αυτό το διάστημα και βρίσκοντας ενωμένε όλες τις φιλευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συντάξουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων και να τον υποβάλουμε στην ε, επόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως. Πρέπει να γίνει αυτό τώρα. Πριν το διορισμό του μελλοντικού ή της μελλοντικής Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδάλλως, θα έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά. Είναι δική μας ευθύνη. Οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις εδώ στο Κοινοβούλιο να τα υποβάλουν αυτά υπόψη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να γίνει τώρα, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν θέλουν μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να γίνει εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καταρχάς να καλωσορίσω τα δύο τρίτα των ε, συμμετεχόντων, των ε, βουλευτών, που είναι η πρώτη τους φορά εδώ. Είναι συγκινημένος, γιατί πριν από 10 χρόνια ε, είχαμε φτάσει να εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτες. είχαμε όμως 7% νέους βουλευτές. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τόσο μεγάλη δημοκρατική έκφραση διασυνοριακά. Θυμηθείτε πώς είναι οι πολίτες που συμμετείχαν στις ευρωεκλογέ την τελευταία φορά για να δημιουργηθεί αυτός ο οίκος της δημοκρατίας, ο διασυνοριακός, σε σχέση με την πρώτη φορά. Εδώ ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης θα αποφασίσουν μαζί να σφυρατήσουν ένα ε, συμβόλαιο αλλαγής αυτό το συμβόλαιο αλλαγή θέλει ουσιαστικά να υποστηριχθεί εδώ από μια ευρεία και σταθερή πλειοψηφία για να αντιμετωπίσουμε τι ε, κατεπίγουσε προκλήσει, τι περιβαλλοντικέ, τι δημοκρατικέ και κοινωνικέ. Θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται προ όφελο όλων. Η συμφωνία αυτή, ένα συμβόλαιο για το μέλλον, θα μπορούσε να ε, επαφιέται στις προσωπικότητες που ε, προέκυψαν ε, απευθεία από τι ευρωεκλογέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα ανώτερα αξιώματα. Χρειάζεται όμω μια αξιόπιστη προσωπικότητα για να τα ενσαρκώνει όλα αυτά, που να υποστηρίζεται από μια ευρεία πλειοψηφία από τι πολιτικέ δυνάμει που νίκησαν στι εκλογέ. Εδώ θα έπρεπε το Συμβούλιο να είχε δεχτεί υπό τον κίνδυνο να υπάρχει στήρα αντιπαράθεση με το Κοινοβούλιο ε, τι προτάσει γιατί αλλιώ θα έβγαιναν όλοι χαμένοι. Σε ένα τέτοιο σενάριο το Κοινοβούλιο θα επιβεβαίωνε τη δυνατότητά του να είναι ο πρώτος ε, δημοκρατικός εκφραστής των Ευρωπαίων πολιτών, των πολιτών της Ένωσης. Και θα είχαμε δώσει απαντήσεις στην δυσφορία σε σχέση με τον κόσμο των πολιτικών. Αυτή θα μπορούσε να ήταν η αρχή η κατάσταση συγγνώμη, στην αρχή της έναρξης της πρώτης συνόδου. Αυτό το σενάριο οδήγησε τους πρασίνους ε, της ομάδας μας να ε, προετοιμάζονται εδώ και μήνες. Γι' αυτό λοιπόν, ε, χωρί επιφυλάξει, εργαστήκαμε σκληρά τι τελευταίε εβδομάδε. Ήταν τεράστια πρόκληση και είχαμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Εκεί όμω ε, που υπάρχει βούληση, μπορεί κανεί να βρει και λύση. Δηλαδή, όποιο θέλει, θέλω σημαίνει και μπορώ. Εδώ όμω εδώ είδαμε τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου επέλεξε ένα δρόμο που θα οδηγήσει οπωσδήποτε στο να γίνουμε εκτελεστέ αποφάσεων που έχουν ληφθεί αλλού, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βεβαίω, η ε, στρατιωτικέ τοποθετήσει πάξου εξεταξιών ε, και εξεβονίμων ε, είναι κάτι που θα γίνει και στην πράξη. Μετά από μια μικροπρεπή ε, διαπραγμάτευση και παζάρεμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε μετά από πέντε μέρε αυτή τη λύση. Όλα αυτά για ένα casting, για ένα διαγωνισμό που δεν πιστεύω ότι με τα αποτέλεσματα που έφερε θα φέρει τι αλλαγέ που περιμένουν οι πολίτε μα και οι κοινωνίε μα. Και άκουσα και θεμητέ ανησυχίε. Ε, πολλοί κατακρίνουν του πρόεδρου αρχηγών και κυβερνήσεων, του πρόεδρου κατών και κυβερνήσεων. Ότι το κοινοβούλιο ως μέρος αυτής της ε, ιστορίας θα πρέπει κυρίως να κατηγορεί τον εαυτό του. Ευχαριστώ για τις επικρίσεις που άκουσα κατά της πολιτικής οικογένειας που εκπροσωπώ εδώ. Αλλά πρέπει να πω στο Συμβούλιο ότι ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεών, μας, των διαπραγματεύσεών σας και εδώ σε μας, η διάθεση να εργαστούμε και εμείς για τους ίδιους στόχους την ερχόμενη πενταετία, δεν φαίνεται να είναι κάτι που το συμμερίζονται όλοι και αυτό δεν είναι καθόλου μια ε, υπερβολική διατύπωση. Οι πολίτε λοιπόν και εμεί ίδιοι δεν υπάρχει περίπτωση παρόλα αυτά να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Εδώ ε, βουλευτέ και συνεργάτε του από του Πρασίνου θα φροντίσουμε να υπάρχει μια Ευρώπη δικαιότερη, βιωσιμότερη και δημοκρατικότερη. Ε, για το κλίμα μα, τη βιοπικιλότητα και του φυσικού μα πόρου. Θέλουμε να είμαστε πρωταθλητέ στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη φορολογική δικαιοσύνη και την οικονομική, καθώ και την ισότητα των φύλων. Η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην εμπροστοφυλακή των ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια δημοκρατία που να είναι πιο συμμετοχική. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων ε, στο επίκεντρο αυτού του πολιτικού ε, βίου και όχι στα περιθώρια. Αυτό το σκοπό, αυτόν τον αγώνα τον άκουσα, το άκουσα να το λέτε πολύ, ότι είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να μονοπολίσει, αλλά πρέπει να το συμμεριστούμε όλοι και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτό πρέπει να γίνει όντω σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σε όλα τα κάτι μέλη, στα ε, δημοκρατικά όργανα, τοπικά, περιφερειακά, ε, ε, σε κάθε επίπεδο. Πολίτε και όλοι μαζί πρέπει να δοθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Συνάδελφοι, λοιπόν, ας μην ε, αυταπατώμεθα. Καίγεται το σπίτι μας. Μπροστά στα κατεπήγοντα της Δημοκρατίας, μόνο ένα τέτοιο συνασπισμό για την κοινοτομία θα μπορέσει να σώσει την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Λάμπερτς, Ο Πρόεδρος Τζάνι, εξ της τη ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Τούσκ, και πάλι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσέφεραν ένα αναξιοπρεπε θέαμα στους πολίτες. Μετά την προκλητική εκστατεία και τις εκλογές της 26 Μαΐου υπήρχε μια ελάχιστη ελπίδα για αλλαγή. Όμως η μέθοδος και τα προγράμματα μας απογοήτευσαν. Το θέαμα που προσφέρθηκε ήταν η θεσμική αντιπαράθεση που παρατάθηκε τις προηγούμενες μέρες. Κάτι που πραγματικά δεν θα κατανοούσαν με τίποτα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Το Συμβούλιο αποφάσισε να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων ε, την ε, μέθοδο ε, που προσπάθησε να προασπιστεί το κοινοβούλιο, αυτή των Spitzenkandidaten, των πρωταγωνιστών υποψηφίων, και τώρα, παρόλο που η μέθοδο θα έφτανε αμφίβολη, παραπονιούνται οι ευρωβουλευτέ για τη συμφωνία που πέτυχαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Λένε ότι δεν με σεβάστηκαν. Μα και εδώ κι εσεί δείχνετε τι υποκριτέ είσαστε. Δεν είσαστε συνεπεί τα λόγια σας, οι πράξεις δεν ακολουθούν τα λόγια σας. Εάν το κοινοβούλιο θέλει να γίνεται σεβαστό, εάν το κοινοβούλιο θέλει πραγματικά να προασπίζεται, ή έστω η πλειοψηφία του κοινοβουλίου θέλει να προασπίζεται την μέθοδο των speech and φροντίστε τα ε, ε, λόγια σας να είναι συνεπή με τις πράξεις σας. Δηλαδή, καταψηφίστε την υποψήφιο που έχει προτείνει το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν το κάνετε αυτό θα μπορούσατε να φανείτε συνεπείς. Ιδάλλως, όπως συχνά έχετε δείξει, όλα αυτά που λέτε φαίνονται λόγια του αέρα. Και δείχνετε ότι ούτε το θεσμικό μα όργανο έχει καμιά αξία, ούτε μπορεί να επηρεάσει τι ευρωπαϊκέ αποφάσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πακέτο του Συμβουλίου, και ας περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις για το πρόγραμμα, διότι ας μην είμαστε προκατελημένοι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν οι βαθιές αλλαγές που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τις ψήφισαν στις 26 Μαΐου. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αλλαγή ρότας που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να επιληθούν τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες και εκεί όπου η πλειοψηφία που έχει κυβερνήσει ως τώρα στην Ευρώπη έχει αποτύχει πλήρω. Η οικονομική κρίση η Ευρώπη σήμερα είναι ήπειρος που αναπτύσσεται με τους βραδύτερους ρυθμούς. Είναι διαρκώς ουραγός. Αυτό είναι αποτέλεσμα των ε, επέσχυντων ε, επιλογών αυτών των θεσμικών οργάνων που δεν βοήθησαν τους πολίτες. Μάλιστα επιβάρυναν ε, την, τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Για την ασφάλεια, εδώ όσοι είμαστε παρόντες από την προηγούμενη θητεία, ζήσαμε δύο μεγάλες και σοβαρότατες απόπειρες σε σχέση με το Κοινοβούλιο και τώρα οι πολίτες μας δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι και ασφαλείς στις πόλεις μας. Δεν αισθάνονται έτσι. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ούτε εδώ βρήκαν μια λύση και απόκριση. Και μετά η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το τρίτο. Δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε προστασία, δεν μπορέσαμε να καλύψουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Αλλά δεν θα το έχουμε πετύχει αυτό εάν ε, δεν προστατεύσουμε τους ίδιους μας πολίτες οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν θα καταφέρουν ποτέ να συμφωνήσουν ποιο έχει δικαίωμα να μπαίνει στην Ευρώπη και ποιο όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πυρός μα μπορεί να ποδοπατηθεί από μεταναστευτικέ ροές και να κατακλειστεί από μεταναστευτικέ ροές που δεν μπορεί κανείς να τι ε, αναχαιτήσει. Για τη δημοκρατία λοιπόν τα ερχόμενα πέντε χρόνια, παρά από το γεγονός ότι η πλειοψηφία ή η πλειοψηφία που θα έρθει ε, δεν κατάφερε να δείξει ότι αυτό το θεσμικό όργανο δεν είναι όργανο δημοκρατικό. Ε, απέκλεισε όσους εκπροσωπούν σχεδόν το 20% των ευρωβουλευτών εδώ μέσα. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε μια θεώρηση της Ευρώπης η οποία είναι ουσιαστικά ελληματική. Ε, και βλέπει μια Ευρώπη χωρίς δικές της δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να ξεκινά από τα εθνικά κράτη, από τις χώρες. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εργάτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, και για όσους λένε ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, there is no way ε, και πρέπει να δίνουμε όλο ένα και περισσότερες εξουσίες στους γραφειοκράτες που ζουν μακριά από τους παλίτες. Λέμε όχι, δεν θέλουμε αυτή την Ευρώπη, ούτε οι πολίτες τη θέλουν. Δεν θέλουμε αυτή την Ευρώπη και αν συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη θα οδηγηθεί, θα οδηγηθεί σε διάλυση οι αποκλήσεις μεταξύ κάτω μελών, των θεσμικών οργάνων δεν θα πετύχουν ποτέ τίποτα. Η δική μας ομάδα ξεκινά από αυτήν την θεώρηση. Μια Ευρώπη όπου τα κράτη-μέλη καθοδηγούν την ευρωπαϊκή συνεργασία, την διαχειρίζονται και προστατεύουν τις διαφορετικότητες που εσείς θέλετε να τις τυποποιήσετε και μάλιστα με νομοθεσία. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τζάνη. Και τώρα για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Λεγκούτκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να σας συγχαρώ να σας ευχηθώ ότι καλύτερο. Νομίζω ότι το πιο προφανές συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από το τελευταίο συμβούλιο είναι ότι το Spitzenkandidat, ο μηχανισμός αυτός των κορυφαίων υποψηφίων είναι ε, παρελθόν, πιο ε, νεκρός και το μεγάλο στο Monty Python, στο σκετσάκι. Και δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι ιδιαίτερα που απήλθε αυτός ο μηχανισμός, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα στις συνθήκες για το Spitzenkandidat, ούτε μία πρόταση, ούτε μία λέξη. Και γνωρίζω φυσικά ότι η στάση πολλών στις ευρωπαϊκές, στην ευρωπαϊκή πολιτική προς τους κανονισμούς και προς τις συνθήκες ήταν αρκετά χαλαρές και αυτό το λέω με ευγενικό τρόπο, ο κύριος Τίμπερμαντς δεν ήταν υποψήφιος των λαών, του ευρωπαϊκού λαού. Ο κύριος Τίμπερμαντς ήταν υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας του πολιτικού σώματος. Και καλά έκανε και έφυγε από το τραπέζι και ελπίζω να μην επιστρέψει κιόλα. Γιατί ουσιαστικά η διαδικασία των επικεφαλής υποψηφίων ήταν να εστιάσουν ε, την εξουσία των πολιτικών ε, οργάνων, όχι να είναι πιο δημοκρατική η πολιτική εξουσία. Το αντίθετο θα έλεγα. Ε, έχουμε λοιπόν πρόβλημα και έχουμε συχνά προβλήματα με τον κανονισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταθερά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Χθε είχαμε πραγματικά ένα λυπηρό θέαμα το οποίο καταδεικνύει πόσο ανοιχτά περιφρονούν πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο το κανόνες. Φυσικά το Συμβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε δικαίωμα να ορίσει τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι η κατάφορη παραβίαση της ε, συνθήκης. Έχει μόνο ε, δικαίωμα να επηρεάσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Το Συμβούλιο φυσικά δεν είναι άμεμπτο αλλά εδώ έχουμε και καλές ειδήσει. Οι καλές ειδήσει είναι σε σχέση με το περασμένο συμβούλιο ότι οι μεγάλες κεφαλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να πετύχουν αυτά που ήθελαν, ήθελαν να επιβάλλουν ουσιαστικά τις δικές τους δομές επί των κρατών μελών με την προσδοκία να γίνονται αποδεκτά όλα αυτά με ταπεινοφροσύνη. Έμα δεν έγιναν αποδεκτά και ελπίζω να διδαχθούν από το πάθημα αυτό και να υπάρξει και μια αλλαγή πρακτικής. Πάνε πια αυτές οι μέρες που δύο-τρεις κυβερνήσεις ε, και οι... οι μέτεροι οι... καθόριζαν την τύχη της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαιτέρως ακούγοντα και τον προηγούμενο μελητή να μιλάει, είναι ότι, κυρίε και κύριοι, δεν φαίνεται να έχετε μάθει από τα τεκτενόμενα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, φαίνεται ότι είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε με την ίδια στρατηγική αλλά ο αριθμό ε, των πολιτών που ανοιχτά επικρίνουν τη στρατηγική αυτή αυξάνεται. Όλο και πιο πολλοί κόσμος επικρίνει τη στρατηγική αυτή τώρα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια για παράδειγμα και είναι σε διαρκή άνοδο ο αριθμό αυτός. Και εσείς φαίνεται ότι κοφεύετε. Αγνοείτε τα σημάδια αυτά, τις ενδείξει προειδοποίηση. και κακώ το κάνετε αυτό γιατί αν δεν αλλάξετε την πορεία σας οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Όπως σας είπα, υπάρχει ε, μία ελαφριά ένδειξη από το τελευταίο Συμβούλιο για μία ενδεχόμενη βελτίωση. Τουλάχιστον εγώ είμαι αισιόδοξο, ήμουν αισιόδοξο. Έχασα λίγο την αισιοδοξία μου όταν άκουσα αυτά που είπατε οι πιο πολλοί εξημών. Όταν έχει γίνει όμως η ζημιά, Μίλτε και μου πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Λεγκούτκο. Πρόεδρε Σίρντεβαν, παρακαλώ εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας Θέλουμε να είστε ένα πρόεδρο για τη διαφάνεια, αμεροληψία και να προασπιστείτε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου έναντι τη Επιτροπή και του Συμβουλίου. Και αυτό με φέρνει στο θέμα που θέλω να θέξω. Το Συμβούλιο και ο πρόεδρο Τούσκ βρήκε μια λύση για το προσωπικό και κάποιοι συνάδελφοι παραπονέθηκαν παρά το γεγονό ότι συμμετείχαν και οι πολιτικέ σα οικογένειε για την επιτεύξη του αποτελέσματο αυτό. Να πω ότι το πραγματικό σκάνδαλο ποιο είναι, ότι τέτοιε λύσει πάντα βρίσκονται και κλεισμένα των θηρών με αδιαφανεί ε, τρόπου. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κοινοβούλιο και έτσι πραγματικά αυτό δεν ανταποκρίνεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη και αυτό προδίδει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ε, καταφέρει ζημιά μεγάλη βλάβη στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ε, μέσα σε εστιατόρια και κλεισμένο των θυρών γίνονται αυτέ τι συζητήσει, λοιπόν. Τι να πιστέψει και ο κόσμο, Ότι το θέμα είναι μόνο οι θέσει. Και όχι το περιεχόμενο. Εμεί ω αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβαμε την εντολή εκατομμυρίων πολιτών εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια αλλαγή, προταστική αλλαγή τη πολιτική. Και αποδεχόμαστε την πρόκληση αυτή. Κάποιοι συνάδελφοι την, τις τελευταίες εβδομάδες ε, έκαναν εντατικές περιπτώδεις διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία συμμαχίας πράσινη, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και συντηρητικοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω το εξή. Πιστεύω ότι οι ελάχιστες συνενέσεις δεν αρκούν για τις ε, πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η αριστερά λοιπόν θέλει αποτελεσματικές λύσεις για την αλλαγή του κλίματος. Χρειαζόμαστε προοδευτικέ ε, πλειοψηφίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα α, κοινωνικά δικαιώματα, να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροδιαφύγη, την φοροαποφυγή. Χρειαζόμαστε λοιπόν και για αυτόν τον σκοπό προοδευτικέ πλειοψηφίε στο Κοινοβούλιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποιο καιρό γιόρτασε τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Θα ήθελα να σας πω ότι για την ομάδα μου είναι πραγματικά παράδεκτο το γεγονός ότι προσυπογράφει αυτή η συμφωνία. Δεν μπορεί να είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπουλά για λίγα ευρώ τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οικολογικά δικαιώματα. Και επίσης έχουμε και τους ακροδεξιούς στην Βραζιλία. Οι πολιτικές αυτές είναι αυτές που δίνουν δύναμη στην ακροδεξία. Αυτό λοιπόν είναι σε αντίθεση με όσα έχουμε συμφωνήσει. Μα κανείς δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Κανείς από τους πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν ε, ζητώ από τους συναδέλφους να τοποθετηθούν σε ό,τι αφορά την ε, ζώνη ελευθερών συναλλαγών και τη σχετική συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Και ναι, η ομάδα της αριστεράς είναι υπέρ μιας ανθρωπιστικής ε, πολιτικής για, την, για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Ε, ο καπτάνιος Καραλάς Αρκέτε, θα θέλαμε να πούμε το εξή. Ας φροντίσουμε να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή της πολιτικής εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και επιτεθειμένοι να τα πράξουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Σίρντεβαν. μην είναι γραμμένοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, έχω στα χέρια μου μια, ένα αντίγραφο τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σα καλώ όλου να το διαβάσετε προσεκτικότατα. Θα ανακαλύψετε πόσε φορέ προδώσαμε τη συνθήκη αυτή. Την προδώσαμε όταν αποφασίσαμε να αφήσουμε μόνο τη στην Ιταλία ω προ την αλληλεγγύη και του μετανάστε. Όταν αποφασίσαμε κατά γράμμα να εφαρμόζουμε του κανόνε για κάποιου, ενώ για κάποιου άλλου κάναμε τα στραβά μάτια, για του φίλου των φίλων δηλαδή. Και εδώ λέτε για διαφάνεια. Αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συνδυάζουν ε, για κλεισμένο των θυρών. Ε, και μετά ε, ενώ λέμε για προστασία του περιβάλλοντο, επιτρέπουμε τη χλυφοζάτη. Ε, ή δεν υπάρχει ελάχιστο μισθό που να ε, εξασφαλίσει τα δικαιώματα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά λέμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Με το προηγούμενο συμβούλιο ουσιαστικά βάλαμε, έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Η ευρωπαϊκή μηχανή έχει πλέον μπλοκάρει πλήρως. Ε, βρίσκεστε σαν καρεκλοκένταυροι ε, ουσιαστικά να κρατιέστε από τις καρέκλες σας, όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βλέπουν τα ίδια προβλήματα να διαιωνίζονται. Πρέπει να αλλάξει κινητήρα αυτή η Ευρώπη λοιπόν. Πρέπει μαζί να αλλάξουμε τους κανόνες. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη εξουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, στην επιλογή των υποψηφίων. Να κάνετε όπως η ε, κυβέρνηση Κόντα και να μην αφήνετε απλώ αυτά που σα προτείνουν ή να τα παίρνετε. Μην γίνεστε πρωταγωνιστέ μια οπερέτα που έχει γράψει κάποιο άλλο. Εμεί είμαστε η φωνή του λαού. Εμείς έχουμε αναλάβει την ευθύνη να υλοποιήσουμε όσα λέει αυτή η συνθήκη. Ας επιστρέψουμε σε αυτά που λέει η συνθήκη λοιπόν. Περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη ανάπτυξη, λιγότερα ε, μαξιλαράκια, λιγότερα ε, γαλλογερμανοί διευθυντέ, λιγότερη ελαζονία. Μαζί μπορούμε να την αλλάξουμε αυτή την Ευρώπη. Μας το ζητούν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Βίντεκομπ. Παρακαλώ, 1,5 λεπτό και για σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή που μιλώ εξ ονόματος της μεγαλύτερης ε, πολιτικής ομάδας εδώ σε αυτό το μέρος. Και θα ήθελα να πω ότι εγώ, αν ε, χρειαζόμουν να πιστώ περαιτέρω ότι το καλύτερο πράγμα για τη Βρετανία είναι να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατόν από εδώ, ήταν ο τρόπος που διεξήχθησαν αυτές οι εκλογές ε, χθε. Γιατί αν ε, έτσι εννοεί αυτό το μέρος τη δημοκρατία, αυτό αποτελεί σοβαρή προδοσία όλων των χωρών που εκπροσωπούνται εδώ. Γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση δημοκρατική διαδικασία αυτή. Και αυτός είναι ένας από τους ε, πολλούς ε, λόγους για τους οποίους η Βρετανία θα πρέπει να φύγει από εδώ. ελπίζουμε μέχρι το Halloween. Και υπάρχει πραγματικά μία επαναλαμβανόμενη ε, ιστορία όπου οι καταπιεσμένοι κατα... καταρρύπτουν και νικούν τους καταπιεστές. Οι Σλάβοι, οι, σκλάβοι, οι α, κύριε Φερχόφστατ, στους χώρες που τους κατέχουν. Και γι' αυτό λοιπόν φεύγει η Βρετανία όπως και να το πούμε και όποιο σύστημα και να χρησιμοποιήσουμε, εμεί θα φύγουμε και χαιρόμαστε που φεύγουμε και εκπροσωπώ την δυτικό και νότιο μέρος του μεγάλη Βρετανία. και από την πρώτη μέρα ήξερα ότι το μέρος αυτός ουσιαστικό ήθελα να αυξήσει τα μέτρα των αλλιέων για να αυξήσει τα εισοδήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν διακόπτει ο Πρόεδρος ε, σε πολλές γλώσσες, λέει η Μρίτρια ότι φεύγουμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου Κατστιάη. Ο κύριος Μαυρίδης, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Right here, Πρόεδρε. Στα συμπεράσματα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η νέα στρατηγική για την επόμενη πενταετία με αφετηρία την προστασία των πολιτών και των ελευθεριών. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προασπίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της όπως αναγνωρίζονται στις συνθήκες και να τους προστατεύει από υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές. ο σεβασμός του κράτους δικαίου λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είναι το μέγιστο συμφέρον και ο ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού μας που μας κρατά ενωμένους απέναντι στις απειλές είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές το ευρωπαϊκό συμβούλιο λοιπόν και η ευρωπαϊκή επιτροπή σήμερα με τον εκπρόσωπό της έβγε αναγνωρίζουν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε και τις παρανομίες και τις απειλές του Ερτογάν στην ανατολική μεσόγειο εναντίον της κυπριακής δημοκρατίας με στοχευμένες κυρώσεις και χωρίς καθυστερήσεις. εκεί κρίνεται το κράτος δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης και σήμερα δηλώνουμε όλοι μας κύπριοι όσοι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Είμαστε από τα ένα μεγάλα από τις μεγάλες ομάδες ε, των Βρετανών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τους φιλελεύθερους, τους πρασίνους, που δεν θέλουμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ άριθμοι αυτή η ομάδα των Βρετανών Ευρωβουλευτών. Και εκείνοι από την πίσω γωνία την αριστερή δεν εκπροσωπούν το σύνολο του Βρετανικού λαού. Σας διαβεβαίω γι' αυτό. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε Τούσκ, για την υπομονή που δείξατε απέναντι στην κυβέρνηση και τη Βουλή μας. Και θα ζητήσω από εσάς και το διάδοχό σας να συνεχίσουν αυτή την πολιτική του χρόνου, της υπομονής και της κατανόησης, ακόμη και όταν φαίνεται ότι η κυβέρνηση μας δεν έχει κανένα σχέδιο Β, ούτε Α ούτε Β. Πάντα το Brexit δεν είναι αναπόφευκτο, γιατί ε, υπάρχει μια μεταστροφή της κοινή γνώμης στο, Ευρω... στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δεν θα βρισκόμασταν εμείς εδώ Υπάρχουν πολλοί από εμά που είμαστε υπέρμαχοι της Ευρώπης, υποστηρίζουμε την Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε και εμείς την υποστήριξη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπυράκη έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Τούσκ, Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Η νέα αρχή που βλέπουμε σήμερα εδώ αποτυπώνει τη νέα συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κέντρου που αποτελείται από το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα τους σοσιαλδημοκράτες τους renew europe και τους πράσινους. μαζί με μια κοινή διακήρυξη κατευθύνσεων οφείλουμε να διασφαλίσουμε στους πολίτες μας πρώτα απ' όλα δουλειές και ανάπτυξη. παρά το γεγονός ότι η ανεργία στην ευρωζώνη κινείται στο 7,5% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία χώρες όπως η ελλάδα χρειάζονται ένα αναπτυξιακό σοκ προκειμένου να προχωρήσουν χρειαζόμαστε δουλειές που θα συνδυάζουν την ψηφιοποίηση της οικονομίας την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μέσω της κυκλικής οικονομίας την εκπαίδευση αλλά και την επανεκπαίδευση. χρειαζόμαστε επίσης να περιφρουρήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας χωρίς εκπτώσεις χωρίς συμβιβασμούς. σε αυτή την πενταετία δεν έχουμε κανένα άλοθη. βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή ξέρουμε το φόβο των ανθρώπων μπροστά στην ψηφιακή μετεξέλιξη ξέρουμε τι συμβαίνει στην ουγγαρία στην πολωνία στη ρουμανία. οφείλουμε να συζητήσουμε να συμφωνήσουμε και να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα διατηρήσει για την ευρώπη τη φήμη ότι είναι η ήπειρος το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς στον πλανήτη. σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Θυμίζω ένα λεπτό ανακεφαλή. Κύριε Γκραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε τους κύριε Σεφτσοβιτς, θα ήθελα να συγχαρώ τους ευρωβουλευτές που επανεκλέγησαν και τους συνεκλεγέντες ε, και να συγχαρώ τον κύριο Τούσκ και για την μακροχρόνια θητεία του, αλλά και γιατί ήταν εκπρόσωπος μιας χώρας Ανατολικής Ευρώπης. Τι παρακαταθήκη θα αφήσετε στο Συμβούλιο, αδιαφάνεια και απόλυτη ανισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μιλώ για τις ηθήνουσες μόνο θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώ και για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στα θεσμικά όργανα. Ούτε εκεί υπάρχει γεωγραφική ισορροπία μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Τι παρακαταθήκη αφήνετε λοιπόν κύριε Τούσκ μία ασυνεπή στρατηγική όσο ό,τι αφορά την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο χώρες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εξακολουθούν να μένουν τιμωρημένε και παραγωνισμένες αποκλεισμένε από το χώρο Σέγγεν. Ενώ είχατε υποσχεθεί στι δύο αυτέ χώρε ότι κάποια μέρα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τα πληρούν, θα ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Εμεί έχουμε ε, εκπληρώσει τι τεχνικέ προδιαγραφέ. Τι άλλη παρακαταθήκη λοιπόν θα αφήσετε, πρόεδρε Τούσκ, τις συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, τις συζητήσεις σε κρυπτό και παραβίστο. Πώς θα πείσουμε έτσι τους Ευρωπαίους πολίτες, τι θα πούμε, πώς θα τους ε, πείσουμε για το ε, ευρωπαϊκό όραμα. Κύριε σας όλοι, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Αλλά έχουμε πραγματικά τιτάνιο έργο μπροστά μας. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάει το Συμβούλιο τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαβουλεύσεις που έχει. Η κυρία ο κύριος, συγγνώμη, Αγγιλάρ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σας όλοι. Πρόεδρε Τούσκ, ε, οι ευρωπαϊκοί πολίτες υπάρχουν, η ευρωπαϊκή θαγένεια υπάρχει, το ακούσατε πολλές φορές. Συνθήκη της Λισαβόνας, χάρτα κοινωνικών, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ε, εδώ και 40 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Και μετά από πολλά χρόνια για πρώτη φορά είχαμε προσέλευση ευρωεκλογέ πάνω από 50%. Και γιατί συνέβη αυτό, γιατί πραγματικά προσελκύσαμε και πάλι τους πολίτες, γιατί είχαν την αίσθηση ότι όταν ψηφίζουν επηρεάζουν τις ηγετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κι όμως πραγματικά καταφέρατε να τα σαρώσετε όλα αυτά. Και δεν μπορέσετε να προσπίσετε ούτε το φραστήμερ μας απέναντι στο βέτο μερικών χωρών που ε, μάλιστα ήταν κατά το τίμερας μόνο και μόνο επειδή ήταν υπέρμαχος του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Επίσης θα πρέπει να προσέξετε τι θα γίνει με τη σύνθεση της Επιτροπής 28 Επιτρόπους και να μην ε, ε, επιλέξετε Επιτρόπους που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές αλλά και τη μεταναστευτική κρίση. Δεν θα πρέπει να ποινικοποιούμε όπως όσους σώζουν ανθρώπινες ζωές όπως συνέβη με την καπετάνισσα του Sea-Watch και θέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να αποφύγουμε επιστροφή σε ε, χώρε που δεν είναι ασφαλεί. Γιατί είχαμε ένα καταβλισμό προσφύγων που βομβαρδίστηκε και μάλιστα είχαμε 40 νεκρού από αυτό το βομβαρδισμό. Θα πρέπει να ε, απαγορεύεται επαναπατρισμό σε τέτοιε επικίνδυνε χώρε. Ευχαριστώ κυρία Νιναγκίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είστε εσεί ο νέο μα πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο καλό νέο που βλέπω από όλα αυτά. Το να πω ότι είμαι απογοητευμένη από την έκβαση του Συμβουλίου θα ήταν πραγματικά εφημισμό. Πρόεδρε Τούσκ, το γνωρίζετε. Ε, δυστυχώς με τις ενέργειες του Συμβουλίου διευρύνθηκε το χάσμα μας από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι πολύ κακό για την δημοκρατία και σίγουρα θα είναι δύσκολο να επαναλάβουμε την προσέλευση την ισχυρή που είχαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Και μάλιστα ε, το Βίσεγκρατ οι πολέμοι του κράτους δικαίου κέρδισαν ε, και αυτή οδήγησε σε χρεοκοπία το Συμβούλιο. Γιατί όλοι είχαμε προσυπογράψει και εσείς και εμείς τη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου και υπαναχωρήσατε. Δεν ε, το ανεχόμαστε αυτό. Πραγματικά αν καταπέσει αυτή η διαδικασία θα δώσουμε το λόγο σε αρνητέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακραίε δυνάμει στο, Ευρωπαϊκό, στο, Ηνωμένο, Συμβουλ... στο Ηνωμένο Βασίλειο συγγνώμη, και αλλού. Θα πρέπει λοιπόν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μη τι άλλο, να στηρίξει τη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου και να, να απορρίψει την απόφαση του Συμβουλίου. Κύριο Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Τούσκ, η επίκρισή μου εναντίον σας είναι για το πακέτο. Το πακέτο δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Είναι αποτέλεσμα μιας ε, ε, πραγματικά θλιβερής διαπραγμάτευσης, ενός παζαρέματος ε, και κλεισμένων θυρών και χωρίς διαφάνεια. Δεν σεβαστήκατε τη διαδικασία μας. Είχαμε υποψηφίου και τώρα αυτή η διαδικασία παραγωνίστηκε τελείως. αλλάξατε τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλοιώσατε τις αρχές μας. Και δεν εκπροσωπείται καν η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όλοι οι συνάδελφοι είναι κατά τη συμφωνία αυτή, αλλά χθε τα ψηφίσατε. Ποιον ξεγελάτε, αν δεν σα αρέσει η συμφωνία, ο κύριο Βέμπερ θα πρέπει να γίνει ε, πρόεδρο τη Επιτροπή ή ο κύριο Τίμερμαν. Και αυτού να ψηφίσετε. Όμω δεν το κάνατε εδώ. Ε, αφήσατε την ε, ε συμφωνία αυτή να περάσει. Αλλαγή στις αξίες μα. Και επίση, κανεί δεν σέβεται το χρόνο. Και όσο για τι διαφορετικέ απόψει που ακούγονται εδώ, μια κυρία πίσω πήρε το λόγο και δεν σα άρεσαν οι απόψει τη και δεν τη σεβαστήκατε. Αν δεν σα αρέσει κάτι που λέει κάποιο, θα πρέπει παρόλα αυτά να κάθεστε και να τον ακούτε. Μιλάτε για δημοκρατία και χθε όλοι σα, χριστιανοδημοκράτε, δεξιά, αριστερή, να ξέρετε όλοι, φροντίσατε να μην εκλεγούν εκπρόσωποι της ID και του CCR. Είναι αυτό δημοκρατία. Τους ε, κλείνετε τι πόρτε. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να πω ότι ο μόνος ε, ύμνο που ε, εδώ αναγνωρίζω είναι ο βουλγαρικό εθνικό ύμνο και σε αυτόν σηκώνομαι προσοχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ε, Κύριε Ευρωβουλευτές, νομίζω ότι αντλήσαμε πολλά σημαντικά διδάγματα τις τελευταίες εβδομάδες. Οι απόπειρε για την καταπάτηση της επιθυμίας και των, ε, της βούλησης του λαού είναι κάτι που έγινε κατάφορα πλέον. Η μεγαλύτερη ομάδα εδώ είναι το ΕΛΚ και θα έπρεπε σωστά να εκπροσωπείται όλες οι συμφωνίες που δεν βασίζονται στις ε, διατάξεις των συνθήκων θα έπρεπε και νομίζω ότι σίγουρα θα συμβεί αυτό να αποτυχάνουν και να απορρίπτονται. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα. Και το τρίτο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να καταπιέζει τις μικρότερες ομάδες στα μικρότερα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χτιστεί μόνο κατά των τεσσάρων του Βίσεγκραντ. Εδώ πρέπει να έχουμε ισχυρά κράτη-μέλη που να είναι σε θέση να συνεργαστούν βάσει των αρχών των συνθήκων. Πρέπει να σεβόμαστε τα συντάγματα της κάθε χώρας. Πρέπει να σεβαστούμε τα θεμέλια και τις αξίες της Υπήρου αυτής. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να φτιάξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Πιστεύω ότι στη διαδικασία αυτή θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Προτείναμε λοιπόν μια δημοκρατική, διαφανή διαδικασία σε ό,τι αφορά την εκλογή του κορυφαίου υποψηφίου. Το Συμβούλιο δεν σεβάστηκε και το ίδιο ισχύει και για τους σοσιαλιστές και για τους πρώην οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με την αρχή την εξή. Το κόμμα, η πολιτική ομάδα που έχει πάρει τις πιο πολλές έντρες στο κοινοβούλιο θα είναι η πολιτική ομάδα που θα επιλέξει το νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συνέβη λοιπόν αυτό. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει τις απόψεις της. Μόνο τότε θα αποφασίσουμε Γιατί το Κοινοβούλιο είναι αυτόνομο πολιτικό όργανο, το μοναδικό άμεσα αιρετό όργανο. Θα λάβουμε λοιπόν τις δικές μας αποφάσεις και δεν πρόκειται να δεχτούμε διταγές από το Συμφούλιο. Είμαι περήφανος που είμαι ε, Βουλγαρός, που είμαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Σημαία και τον Ευρωπαϊκό Ύμνο. Αυτά θα πρέπει να μας ενώσουν σε ό,τι αφορά μια ασφαλή ευρωπαϊκή πατρίδα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Τούσκ, όντως το Συμβούλιο ολοκληρώθηκε. Ε, διαβάσαμε τα αποτελέσματα, είδαμε την πορεία των διαπραγματεύσεων και δεν ήταν πολύ ευτυχής όλες αυτές οι εξελίξεις. Πάνω όμως από όλα θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από όλα αυτά. Και σίγουρα πολλά μπορούν να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το δίδαγμα και πολλά να βελτιωθούν. Γιατί περιμένουμε ε, από ο κόσμος περιμένει από εμά, έχει δείξει την εμπιστοσύνη του και περιμένει από εμά να υποβάλουμε ένα πρόγραμμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις των καιρών. Δεν έχουμε πια χρόνο να μιλούμε για τον καταμερισμό των θόκων και των αξιωμάτων, να πούμε τι συγκεκριμένα θα κάνουμε την επόμενη πενταετία. Και επίσης να λογοδοτήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην μείνουμε πίσω, να μην μείνουμε ουραγοί της Αμερικής ή της Κίνας, αλλά να είμαστε ηγέτες η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίων. Να σταματήσετε πια την κατανομή των θόκων. Μιλάτε για συγκεκριμένα αποτελέσματα και επικεντρωθείτε στην υλοποίησή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε ε, Τούσκ, κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Σεφτσοβίτση. θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά, οι πολιτικές ομάδες ε, επέμειναν, επέμειναν προκειμένου να τηρηθεί η αρχή των Spitzenkandidat. Δεν το καταφέραμε. Γιατί τελικά και κλεισμένο των θυρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ελήφθησαν αποφάσεις. Μιλάμε για γεωγραφική ισορροπία, η οποία επίσης δεν έγινε σεβαστή όμως. Και τελικά θύματα είναι οι χώρες ε, του Βίσεγκραντ, που είχαν ένα καλό υποψήφιο, ο οποίο είναι εδώ μεταξύ μας, στην Ολομέλεια. Και αν όντω ο, ο υποψήφιος δεν εκλέχθηκε μόνο και μόνο επειδή είναι από την περιοχή αυτή, από την περιφέρεια αυτή, αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ κακό σημάδι, μια κακή ένδειξη για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και την επικοινωνία με τους πολίτες, γιατί δεν θα πιστεύουν αλλιώ στην συμμετοχική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Μαριάννη. Μαριάννη. Le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τους νεοεκλεγέντες ε, που έχουν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη με, κάποιες, ε, ε, με κάποια οράματα και ψευδεστήσεις. Άκουσα ωραίους λόγους για τη δημοκρατία, για την αρχή του σεβασμού των μειονοτήτων, αλλά ωραία τα λόγια, τα έργα που είναι, τα συγκεκριμένα τα αυτά αποτελέσματα. Χθε ε, μείναμε πολύ στον αποκλεισμό ε, ευρωβουλευτών που αντιπροσωπεύουν το 20% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε είναι από το ECR, είτε είναι από την ομάδα ID ε, και εμείς ε, έχουμε κατά νου Ευρώπη. Ίσως δεν συμπίπτει με τη δική σας ιδέα για την Ευρώπη. Είναι ωραία να ε, προασπίζουμε τις ε, τις αρχές, αλλά θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλα. Χθε έγιναν κάποιες συμφωνίες μεταξύ μετέρων για να αποκλειστούν 20% των ευρωβουλευτών και μάλιστα θα περιμένουμε χωρίς πολλές ψευδοστήσεις και την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να ε, αποκλείσουμε πάλι το 20% των ευρωβουλευτών στην κατανομή των ε, θέσεων μελών στις διάφορες επιτροπές. Γιατί αν συμβεί και αυτός ο αποκλεισμός θα, δω, θα καταλάβω ότι είναι μόνο θεωρία αυτή η προσήλωσή σας στις αρχές και τις αξίες. Ο κύριος Όλεγκας, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ στην Ολομέλεια, να σα συγχαρώ για την εκλογή σα στη θέση του Προέδρου και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Τούσκ και τον Αντιπρόεδρο Σεύτσοβιτ για την ομιλία που μα απέφτυναν. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για την απουσία ισορροπία εκπροσώπηση μεταξύ Ανατολή και Δύση στις κορυφαίε αυτές θέσεις. Θα έπρεπε να συζητάμε το πώς οι εκλεγμένοι βουλευτές θα έπρεπε να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τα αξιώματα αυτά και το πώς θα συνεργαστούν και θα έπρεπε να συνεργαστούν τα δύο θεσμικά όργανα. Αν δεν πετύχουμε να την ίση εκπροσώπηση, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε και τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες η δημοκρατία, η πρόκληση της αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά, συνάδελφοι, επιτάσσουν κοινέ αποφάσεις. Για να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους μας θα πρέπει να πετύχουμε καλύτερη τη θεσμική συνεργασία και βλέπουμε ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να μας δείξει κάτι τέτοιο σήμερα. Εμείς όμως καλούμε το Συμβούλιο να το κάνει αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα για την απάντησή του εκ μέρους της Ευρωπαϊκής ο κύριος Εύκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους βουλευτές, γιατί απέδειξαν ξεκάθαρα ότι ήρθαν ανανεωμένοι με φορτωμένες μπαταρίες και υψηλές φιλοδοξίες για την ερχόμενη θητεία. Από όλε τι παρεμβάσει άκουσα ξεκάθαρα ότι υπάρχει σύγκληση. Σύγκληση μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων για μια στρατηγική ατζέντα για το μέλλον. Εργαζόμαστε σκληρά τα τελευταία πέντε χρόνια για να βεβαιωθούμε ότι, ο Ευρωπαϊκό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παραμένει μόνο πρωταγωνιστή στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά ότι παραμένουμε και η πρώτη βιωσιμότερη οικονομία στον κόσμο. Ε, μια από τι μεγαλύτερε λοιπόν ευθύνε όλων μα σε αυτή τη νέα θητεία είναι να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τη σωστή εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Νομίζω ότι αυτό που είπαν ο κύριος Τσόρος, ο κύριος Πόνς, η κυρία Γκαρσία Πέρες, ε, ο κύριος Λάμπερτς, ότι πρέπει δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια τα αξιοποιούμε για μια κοινωνικότερη, πρασινότερη και δικαιότερη Ευρώπη. Να το θυμόμαστε όλοι σε κάθε επόμενο βήμα μας, όταν θα σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας και τις δουλειές μας για το μέλλον. Ε, θα συμφωνήσω με τον αγώνα που οι περισσότεροι είπατε ότι θέλετε να δώσουμε. Η οικονομία μας να παραμείνει πρώτη, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ένδυα. Ο καθένας να μπορεί να δει ότι έχει κάποιο μέλλον στα πλαίσια αυτής της νέας οικονομίας τις βασικές ε, κεντρικότερες περιοχές ε, του σήμερα ή τις πόλεις και τα σπίτια που καταναλώνουν πολλή ενέργεια και χτίστηκαν πριν από πολλές δεκαετίες στις μεγάλες πόλεις. Πρέπει να δώσουμε νέες ελπίδες, νέες προοπτικές ε, για το μέλλον στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος. Κάτι που επίσης τονίστηκε παρελειμμένος, κάτι που είπε η κυρία Γκαρσία Πέρες, ότι πρέπει να έχουμε χειροπιαστά μέτρα, αλλά θα πρέπει να ληφθούν και σχετικές αποφάσεις για το ερχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο, δεν μπορούμε να χάνουμε εβδομάδες, μήνες και ώρες ε, ατελείωτες με ένα πρόγραμμα που απλώς μένει στα χαρτιά όσο δεν υπάρχει οικονομική στήριξη για αυτό χωρίς στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να γίνει συμφωνία Πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος για την ε, επιτυχή ε, εξέταση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Χρειαζόμαστε μια οικονομία που ανοιχτά θα είναι και πράσινη και καθαρή και ανταγωνιστική είναι σαφέ σε σχέση με όσα κάναμε ήδη ότι αυτή τη φιλόδοξη προσέγγιση τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τι τεράστιε ε, μεγάλε ανάγκε. Την ε, ρομποτοποίηση, την ψηφιοποίηση, την καθαρή ενέργεια ε, και για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον ανταγωνισμό τη Κίνα. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στου πολίτε, στο περιβάλλον, στι διεθνεί συνθήκε, του κανόνε και τι υποχρεώσει μα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω στον κύριο Σίρντεβαν ότι ό,τι νέε εμπορικέ συμφωνίε υπάρξουν θα συζητήσουμε και μαζί σα. Και όλε να είστε βέβαιοι ότι θα σέβονται τα υψηλότερα, πρότυπα, ε, τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στα περιβαλλοντικά, τα εργασιακά, την οικονομία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή μα απάντηση στι τάσει προστατευτισμού που είδαμε να αναδύονται ανά τον κόσμο από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω θα σα εξηγήσουμε την κάθε διαδικασία βήμα-βήμα και την κάθε φιλοσοφία την, κάθε, την όλη φιλοσοφία που υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις συμφωνίες. Συνάδελφοι, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι για όσους φεύγετε θα λυπηθούμε που θα αποχωρήσετε, ειδικά αυτό να το πω στους Βρετανούς. Ε, και σε όσους βρίσκονται τα δέντρανα πιο ψηλά, θα πω με όλη τη διπλωματική τέχνη που διαθέτω ότι δεν θα δεχτούμε μαθήματα ε, διακυβέρνηση και διαχείριση των πραγμάτων από εσά. Πρόεδρε του Ευρωκοινοβουλίου λοιπόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήθελα να ολοκληρώσω την πρώτη μου ομιλία εδώ στο Κοινοβούλιο λέγοντας ότι θα ας βεβαιωθούμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα τα αξιοποιήσουμε και ότι ότι η πενταετία αυτή θα είναι όσο δυνατόν ευρωπαϊκότερη, διότι ο κόσμος χρειάζεται μια ενωμένη, ισχυρή και ε, εύρωστη Ευρώπη. Ευχαριστούμε και τώρα η απάντηση του Πρόεδρου Τούσκ. Παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ να έχουμε αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σήμερα θα αποφύγω οποιοδήποτε σχόλιο επ' αυτού. Ελπίζω οι νέοι ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι ε, οι νέοι θύνοντες να δείξουν ισορροπία από κάθε άποψη. Μάλιστα, ευχαριστώ τον πρόεδρο Τούσκ, τον αντιπρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Σεφτσοβιτς ε, που ήρθαν σήμερα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση και να σας ε, προτείνω κατά απόκληση από το άρθρο 202 ε, να εγκρίνουμε αμέσως τα πρακτικά της χθεσινής συνόδου και ε, τα υπόλοιπα πρακτικά θα υποβληθούν για έγκριση στην έναρξη επόμενη συνόδου. Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσει. Οι σοσιαλιστικοί δημοκράτε πρότειναν τα εξή για τι τροποποιήσει στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Η κυρία Κοταγιάρα αντικαθιστά την κυρία Μύρια Μντάλη στην Επιτροπή ε, Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια και ο ο κύριο Κοζολίνο αντικαθιστά τον κύριο Πιτσαπία στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν παρατηρήσει για αυτέ τι αντικαταστάσει. Ε, από ό,τι φαίνεται όχι. Οπότε εγκρίνονται οι σχετικοί διορισμοί. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνεργασία και κηρύξω την διακοπή της Συνόδου Ολομέλειας. Λύεται η συνεδρία.